Good afternoon, colleagues, uh, for a next uh, Ευχαριστώ. Στην συνεδρίαση της ΕΚΟΝ έχουμε μια πολύ σύντομη ανακοίνωση από πλευράς Προεδρού. Θα υπάρξει μια ανοιχτή συνάντηση συντονιστών την 1η Μαρτίου από 12 μέχρι 1.30. και Θα έχετε τη δυνατότητα να ανταλλάξετε απόψεις και με την αρμόδια της αρχής για την... This meeting will also be uh, Την αρχή για την εκαθάριση των πιστοτικών ιδρυμάτων. Έχουμε τρία θέματα, καταρχάς μικρομεσαίες, μετά έχουμε ε, τους εμπορευομένους ε, ε, πρώτες ύλες και βασικά εμπορεύματα, αλλά θα ξεκινήσω με τον κύριο Κάρας, για την πρόσβαση ε, των μικρομεσαίων στις πηγές χρηματοδότησης. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που σε μια έκθεση για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ασχολούμαστε με τέτοια θέματα. Και είναι εδώ και ο συνάδελφος, ο οποίος την τελευταία φορά ήταν συντάκτης της έκθεσης της σχετικής. Να σας παρουσιάσω ποια είναι τα σημεία κλειδί της ε, έκθεσης αυτής, του σχεδίου αυτού έκθεσης. Είναι σαφές ότι όλα τα μεγάλα σχέδια των τελευταίων ε, χρόνων ο σκοπό είχαν να ενισχύσουν τον τομέα των μικροπεσαίων επιχειρήσεων και το Εύση και τα υπόλοιπα όλα τα προγράμματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν εξακολουθούν να είναι ο καθοριστικός κρίκος στην ευρωπαϊκή αγορά για την ανάπτυξη της επενδύσεις και της θέσης απασχόλησης. Και ως εκ τούτου θα πρέπει στο μέλλον να εξασφαλίσουμε να σκεφτόμαστε σε κάθε νομοθεσία ποιε θα είναι οι συνέπειε για την πραγματική νομοθεσία, για πραγματική οικονομία. Και συνέχεια, πάντα απαιτούσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει υπόψη το Better Regulation, τι καλύτερε ρυθμίσει, αλλά και το Small Business Act και σε αυτά πάντα να τονίζει και να κοιτάει ποιε θα είναι οι συνέπειε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και εδώ λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την ΕΣΜΑ και το SSM να παρακολουθεί επακριβώς τις νομοθετικές εξελίξεις. Γιατί όλο και πιο συχνά τι βλέπουμε. Ότι με τις ε, πράξεις κατά και με τις ρυθμίσεις, ε, τις εποπτικές, συχνά πρώτα ρυθμίζεται το θέμα των πολιτικών ε, και των οπτικών αποφάσεων και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και αντιφάσεις, μη σας πω και εκ παραλλήλου θα πρέπει να φροντίσουμε για την ε, ποικιλία και τη διαφορετικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό το φαινόμενο και να το λάβουμε υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται διάφορες ε, μορφές χρηματοδότησης οι μικρομεσαίες σε όλες τις φάσεις του κύκλου εργασιών τους, από τις ε, startups, τις νεοφυείς, μέχρι και την μεταβίβαση τέτοιων επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένα και στα μέτρα τους ε, μέτρα χρηματοδότηση. Ένα λοιπόν στοιχείο τη έκθεση είναι το εξή. Τον ε, παράγοντα της υποστήριξη, τον οποίο τον είχαμε εισαγάγει ήδη στη Βασίλεια 2 να τον ε, επιμηκύνουμε. Σε ό,τι αφορά όλε τι μορφέ χρηματοδότηση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα κλασικά δάνεια των τραπεζών θα αποτελούν και στο μέλλον το κλασικό τρόπο χρηματοδότησης των μικρομεσαίων. Αλλά παράλληλα αυτά θα υπάρχει η αγορά ε, η κεφαλαιοχική. Δεν θα πρέπει να παρέσουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια υγιή, ένα υγιή και σωστό τραπεζικό τομέα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και ένα από τα βασικά μέτρα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη χορήγηση δανείων είναι ακριβώς η επιμήκυνση, η παράταση του παράγοντα supporting αυτό των υποστηρίξη. Δεν προκάλεσαν οι σε την κρίση, αλλά αυτές είναι που πλήττονται πιο πολύ από κάθε άλλη εταιρεία. Και γι' αυτό αυτός ο supporting factor αποτελεί ένα από τα πιο απαραίτητα και δίκαια μέτρα για να ελαφρύνουμε τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και την δυνατότητα να καταστεί μόνιμο μέτρο αυτό ο φορέας, αυτός ο παράγοντας και να χρησιμοποιείται ανα πάσα στιγμή. Και γι' αυτό είναι σημαντικό επίσης να μην υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του Better Regulation, το θέμα της αναλογικότητας και εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, να υπάρχει ένας επακριβής ορισμός του όρου. Χρειαζόμαστε εναλλακτικέ επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ε, μικρομεσαίες, πέρα από τη χορήγηση πιστώσεων δανείων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει μια ευρωπαϊκή κουλτούρα για την ανάληψη κινδύνου και για την ε, κεφαλαία αγορά. Θα πρέπει να αναπτυχθεί λοιπόν μια τέτοια κουλτούρα. Και γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντική αυτή η συζήτηση και η συζήτηση για την Κεφαλική, την κεφαλική Ένωση. Και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες ε, ε, τράπεζες είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και έχουν πολύ σημαντική θέση. Και σημείο κλειδί είναι το τι γίνεται με τους νέους ανθρώπους και με τις νέες επιχειρήσεις. Μόνο όποιος έχει την απαραίτητη οικονομική βάση μπορεί να αναλάβει ρίσκο και να πειραματιστεί και με εναλλακτικέ μορφές χρηματοδότησης. Και το πόσο σημαντικό είναι αυτό ποιος ε, νέος ε, επιχειρηματίας ε, ξέρει ποιες είναι ακριβώς οι υποχρεώσεις της τράπεζας σε περίπτωση που απορρίψει ε, την, πρόταση, την αίτηση δανείου. Όλες αυτές τις γνώσεις λοιπόν θα πρέπει να τις διαβιβάσουμε στους νέους επιχειρηματίες γιατί έτσι μόνο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και επίσης ε, το κόστος της πρόσβασης στις κεφαλαίες αγορές θα πρέπει να μειωθεί μόνο με μια διαφάνεια σε ό,τι αφορά την αναφορά των υποχρεωτικών εξόδων μπορούμε να εγγυηθούμε καλύτερη συμμετοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι περνάμε στις startups, στις νεοφύης επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτές ε, πρέπει να πούμε ότι τις επόμενα χρόνια θα είναι ιδιαίτερη σημασία. Από αυτέ εξαρτώμαστε για να κρατήσουμε τι καλύτερε ιδέε και τα καλύτερα κεφάλια, αν θέλετε. Γιατί οι Γάλλοι θα διαφύγουν το 2014 στην Ασία συλλέξηκαν πιο πολλά μέσα και κονδύλια για το crowdfunding στην Ασία παρά στην Ευρώπη. Θα πρέπει από νομοθετική άποψη λοιπόν να ε, αντισταθμίσουμε την κατάσταση. Και εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι είναι διαφορετικέ οι συνθήκε που επικρατούν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την υπηρετική Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, και για το P2P και για το crowdfunding χρειαζόμαστε ενιαία νομοθεσία και για τις υπόλοιπες ε, νέες μορφές ε, χρηματοδότησης και για τις νεοφύης επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν πλήρη επισκόπηση της αγοράς εργασίας στη χώρα τους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε κάθε χώρα ισχύουν διαφορετικέ προδιαγραφέ. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν η διαμόρφωση τη νομοθεσία. Χρειαζόμαστε ίδιε συνθήκε πλαίσιο, ίδιου όρου πλαίσιο. Και αν έχουν όλα τα κρατημέλη One Stop Shop μέσα του οποίου μπορούν να ενημερωθούν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να κάνουν τα απαραίτητα βήματα από ένα κεντρικό σημείο για τις σχετικές αιτήσει τους. Και ελπίζω και στο σημείο αυτό να μάθουμε με τα One Stop Shop ε, να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να καταλάβουμε ότι είναι υπερβολικός ο κετοματισμός που επικρατεί στην παρούσα φάση. και ότι δεν ε, εκμεταλλευόμαστε πλήρω τι ευκαιρίε και τι δυνατότητε που έχουμε. Μόνο λοιπόν αν συμβεί κάτι τέτοιο. Και τελικά μπορεί κανεί από τη Μαντρίτη στο Ταλίν, στο Βουκαρέστι να έχει τι ίδιου όρου, τότε μόνο θα υπάρχει πραγματικό συμφέρον να μείνει κανεί με την επιχείρηση στην Ευρώπη και να μην μετακατασταθεί κάπου αλλού στον κόσμο. Και έχω πολλά παραδείγματα να σα δώσω όπου παράγεται το λογισμικό μεν στην Ευρώπη, αλλά μετά φεύγει. Γιατί οι δυνατότητε χρηματοδότηση για την εφαρμογή του IT δεν ε, υφίστανται. Αυτά όλα βλάπτουν, βλάπτουν την οικονομία. Προσπάθησα λοιπόν ε, με το μορφότυπο που επιβάλλεται, γιατί είναι έκθεση πρωτοβουλία, καταλαβαίνετε. Προσπάθησα λοιπόν να θίξω όλα αυτά τα στοιχεία. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεπεράσουμε και να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία με τις τροπολογίες που θα κατατεθούν και καλώ όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή προκειμένου μέχρι τέλη Ιουνίου τελικά να έχουμε προετοιμάσει μια εξαιρετική έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης τους. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάρας για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ζήμων. Thank you. And, uh, Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και προς τον εισηγητή. Ιδιαίτερα διαφωτιστική η παρουσίαση του, πλήρης παρουσίαση, πάνω σε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει τίποτα στην έκθεση που εμείς στην σοσιαλιστική ομάδα θα λέγαμε ότι διαφωνούμε. Νομίζω ότι περιλαμβάνονται κοινά μεταξύ μας στοιχεία, έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες και ίσως ε, τελικά να διαφέρουμε τα μικρά γράμματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια κάποια κίνη αντίληψη. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο τώρα για κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες θα θέλαμε κι εμείς ε, να προσθέσουμε κάποια επιμέρους στοιχεία. Αλλά πριν από αυτό να κάνω μια γενική παρατήρηση. Η έκθεση είναι σαφής σχετικά με την κεντρική, ε, τον κεντρικό ρόλο της χρηματοδότησης από πλευράς των τραπεζών. Και αυτό πάντα ίσχυε. Οι τράπεζες είχαν πάντα κεντρική, κεντρικό ρόλο να παίξουν. Παρ' όλα αυτά, η δική μου εμπλοκή σε τέτοιου είδους ε, συζητήσεις χρηματοπιστωτικές κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Και για όλα αυτά τα χρόνια φοβάμαι ότι η συζήτηση δεν αλλάζει ποτέ. Για ένα κοινό μόνιμο πρόβλημα. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων τέτοιου μεγέθους η οποία δεν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα, να μην πω δεν έχει βελτιωθεί καθόλου στις ε, μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες ε, και ε, στο δικό μας πλαίσιο το οικονομικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι έκαναν πολλά, έγιναν πολλά σε υψηλό επίπεδο αλλά νομίζω ότι απέδειξε ο τρόπος με τον οποίο προσπαθήσαμε μέχρι τώρα ότι δεν ήταν αποδοτικός. Αυτό το οποίο λοιπόν καλούμεθα τώρα πια να κάνουμε, όσο και αν ακούγεται κάπως ερετικό, θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το οποίο λείπει από τις μορφές χρηματοδότησης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θέλω τώρα να περάσω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν κάποια κενά στη χρηματοδότηση και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους δεν έχει νόημα πολλές φορές, οικονομικό νόημα, να δανείζουν σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πλέον σαφές. Και γι' αυτό να προσπαθήσουμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους μόχλευσης και έβρεσης γενικότερα μορφών χρηματοδότησης. Οι μικροχρηματοδοτήσεις, οι μικροπιστώσεις, ίσως εδώ να έρχεται σε επαφή με το πιστοτικό κομμάτι των τραπεζών, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε κάποια προγράμματα δανειοδότησης μέσω των οποίων το κράτος δανείζει τις τράπεζες για να δανείσουν τις μικρομεσαίες. Αυτό δεν ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα πρέπει να δούμε αυτά τα συστήματα αν δουλεύουν καλά και αν μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Ίσως να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες να χρηματοδοτηθούν και σε επίπεδο ανάπτυξης τους χρησιμοποιώντας φυσικά και τις κεντρικές ευρωπαϊκές δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και χώρες, θυμίζω, στις οποίες αυτό το οποίο είπα ότι ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ισχύει και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις με τις κρατικές χρηματοδοτήσεις γιατί επαναλαμβάνω ότι τα μεγάλα πιστοτικά ιδρύματα δεν θεωρούν ιδιαίτερα ελκυστική τη δραστηριότητα δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης θέματα αμοιβαίας χρηματοδότησης, μικροχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ε, τα λεγόμενα business angels, οι άγγελοι της επιχειρηματικότητας. Άτυπες θα έλεγε κανένας ή έκτακτες μορφές χρηματοδότησης. Αυτά είναι τομείς τους οποίους θα πρέπει να ασχοληθούμε, με τους οποίους θα πρέπει να ασχοληθούμε Για τις τράπεζες τώρα θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των μικρομεσαίων για τις δυνατότητες των πιστοτικών ιδρυμάτων και θα υπάρξει επίσης και πρέπει να υπάρξει και καλύτερη εφαρμογή των μέσων χρηματοδότησης και των διαδικασιών καλύτερα, τα λεγόμενα one-stop shop. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το ρόλο μας σαν κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια γενικά πρέπει να παρεύουν στο συγκεκριμένο τομέα έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένων εταίρων στο επίπεδο της χρηματοδότησης. Η ίδια η αγορά δεν πρόκειται να καταστήσει το σύστημα πιο δίκαιο, οπότε εμείς πρέπει να, είμαθε, να παρόντες. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισήγητη. για μια εξαιρετική προσπάθεια. Νομίζω ότι μπορούμε να συνασπιστούμε πίσω του και να μπορέσουμε να προωθήσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος των συντηρητικών δεν είναι παρόν και γι' αυτό θα διαβάσω τη δήλωσή του. Θέλει να ευχαριστήσει τον κύριο Καράς για την προσπάθεια την οποία έκανε. Πιστεύει ότι πολλές από τις ιδέες στην έκθεση είναι πάρα πολύ καλές και θα τις συνυπογράψει. Έχει όμως και ορισμένες παρατηρήσεις να κάνει. Uh, paradoxically, uh, to all the efforts uh, we put in simplify regulatory... Θα πρέπει να απλοποιηθεί το διακανονιστικό πλαίσιο το ισχύων για τις μικρομεσαίες. Όταν παράγουμε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις καθιστούμε το περιβάλλον πολύ πιο δύσκολο για τις μικρομεσαίες. Απαιτείται μεγαλύτερη λοιπόν διακανονιστική ελευθερία, μεγαλύτερη ευελιξία, Πολλές φορές ε, απουσία επιβάλλεται ρυθμίσεων και κανόνων. Αυτό είναι ευεργετικό για τις μικρομεσαίες, θα επιταχύνει την ανάπτυξή τους, θα διευκολύνει τις ε, νέες επιχειρήσεις, την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τις λεγόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις. Και έχει σημασία για τις μικρομεσαίες να μπορούν να την χάνουν και φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων μερικές φορές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και έτσι θα υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν και αυτά με τη σειρά τους, με τη δική τους εθνική προοπτική τα προβλήματα που έχουν οι μικρομεσαίες και γι' αυτό θεωρούμε ότι η περαιτέρω εναρμόνιση του νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αποτελέσει τροχοπέδι στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Πέραν τούτου, ο κύριος Σόλτσοκ θα υποβάλει μια σειρά από τροπολογίες σε κάποιες από τις παραγράφους. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα στις παραγράφους 23 και 24 για την περαιτέρω εναρμόνιση την οποία εσείς προτείνετε. Ο κύριος Σόλτσοκ θεωρεί ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τις προτάσεις σας ιδιαίτερα σε σχέση με τα λεγόμενα crowdfunding, τις συλλογικές χρηματοδοτήσεις μέσω διαδικτύου. Ο κ. Σόλτσοκ υπογραμμίζει επίσης τη σημασία που έχουν οι φορολογικές απαλλαγές για τις μικρομεσαίες. Στις παραγράφους 9 και 10 λέγει ο κ. Σόλτσοκ ότι θα ήθελε να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή των εναλλακτικών χρηματοδοτικών μεθόδων, όχι μόνο τράπεζες δηλαδή λέγοντας όμως ότι φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον ρόλο των τραπεζών στη χρηματοδότηση. Τώρα για την παράγραφο 20 συμφωνεί ότι θα πρέπει να αξικολογήσουμε το υπάρχον διακανονιστικό πλαίσιο με διαφορετικό τρόπο και υπογραμμίζει την ανάγκη να το κάνουμε αυτό από πρακτικής επόψεως και να προσπαθήσουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει μια τέτοια προσπάθεια σε επίπεδο κρατών μελών. Και επίσης προτείνει τροπολογίες στην παράγραφο 7 για, τον, για την απομάκρυνση των μη απαραίτητων εμποδίων για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων. Πάντως η πρότασή σας είναι μια καλή βάση και ελπίζουμε μέσω και των τροπολογιών μας θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση και να εξετάσουμε και τις υπόλοιπες τροπολογίες. Αυτά από πλευράς του κυρίου Όζοκ. Ο κύριο Τεμπάκερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και από δική μου πλευρά να ευχαριστήσω καταρχά τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεση, το οποίο όντω περιλαμβάνει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Πολύ ενδιαφέρουσε κάποιε παράγραφοι και ήμουν όντω ε, εισηγητή τη τελευταία έκθεση ίδια πρωτοβουλία που καταπτύχθηκε από την Επιτροπή μα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Και νομίζω ότι κοιτώντα το πώ έχει η τρέχουσα έκθεση, σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε την ε, παλιά έκθεση, γιατί πολλέ συστάσει κάναμε ω Κοινοβούλιο και ω Επιτροπή τότε προ την Κομισιόν. Και θα πρέπει να δοθεί ένα follow-up. Ίσως από εκεί λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ένα σχέδιο δράση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι τμήματα του σχεδίου δράση ε, έχουν εφαρμοστεί, λειτουργήσαν, ποια θα πρέπει να ενημερωθούν, και ποια θα πρέπει να έχουν κάποια συνέχεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Ένα δεύτερο σχόλιο. Η έκθεση θέτει μεγάλη έμφαση σε ό,τι αφορά τις ε, τραπεζικά δάνεια. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ αυτό σημαντικό για την οικονομία, αλλά σε καιρούς ε, κρίσης ζητούμε από τις τράπεζες να έχουν μικρότερους ισολογισμούς, να αναλαμβάνουν λιγότερους ε, ε, λιγότερα ρίσκα και φυσικά παντού υπάρχει credit crunch. Και σε κάποια κράτη-μέλη βλέπουμε όμως ότι λίγο πολύ τα δάνεια έχουν παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, αλλά έχουν γίνει πιο αυστηροί οι όροι χορήγηση των δανείων. Και αυτά τα στοιχεία λοιπόν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι καλός και άγιος ο τραπεζικός τομέας σε ό,τι αφορά τα δάνεια και σε ό,τι αφορά τους περιοριστικούς όρους για τη χορήγηση των δανείων, αλλά σημαντικό είναι να κοιτάξουμε και μία διαφοροποίηση, μία ποικιλία να υπάρχει στο σύστημα. Γιατί και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει από το one size fits all. Δεν μπορεί να υπάρχει μία λύση για όλε. Μιλάμε για νεοφυεί, μικρέ, ε, ε, venture capital, μικρομεσαίε επιχειρήσει, μικρέ με 4-5 άτομα μέχρι και επιχειρήσει με εκατοντάδε άτομα. Είναι μεγάλη η διαφοροποίηση. Θα πρέπει να λεφτεί λοιπόν αυτό υπόψη σε ό,τι αφορά τι συστάσει που θα κάνουμε και ενδεχομένω λοιπόν να πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ το όλο σύστημα που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των μικρών μέσων επιχειρήσεων. Χρειάζεται λοιπόν να μπορούμε να αναλάβουμε και λίγο παραπάνω κίνδυνο, μεγαλύτερη καινοτομία, να ε, προκριθούν και νέε μορφέ χρηματοδότηση και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφερθούν όλα αυτά στην έκθεση. Συνολικά. Πιστεύω λοιπόν ότι πολλά είναι τα καλά και θετικά στοιχεία τη έκθεση, αλλά και εγώ θα προσπαθήσω να προσθέσω κάποιε ιδέε από, τις, από αυτές τις οποίες μόλις σας παρουσίασα και φυσικά να υπάρξει και ένα follow-up από την προηγούμενη έκθεσή μου, να δούμε τι ε, πήγε καλά, τι δεν εφαρμόστηκε και τι μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει καλύτερα από ό,τι κάνει έως σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντεμπάκαρ και τώρα από πλευράς της ΓΚΟΕ Παλώμα Λόπες Ερμέχο. Muchas gracias, Presidente. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα από τα σημεία της έκθεσης, εκεί όπου αναγνωρίζει ότι τα τραπεζικά δάνεια είναι παραδοσιακά η πιο σημαντική πηγή ε, χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπογραμμίζεται ο ε, σημαντικός ε, ρόλος των ε, τραπεζών που έχουν συγκεκριμένη τοπικό, συγκεκριμένο τοπικό χαρακτήρα και έχουν και πολύ στενότερη σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά κάποιο τρόπο αναγνωρίζει πως οι πολιτικές της Κομισιόν ε, προχωρούν εις βάρος των όσων ήταν παλιότερα το πρότυπο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θέλω να με σαφή. Τα προβλήματα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων δεν είναι πρόβλημα του μοντέλου πίστοσης είναι αποτέλεσμα της τραπεζικής συγκέντρωσης και των επιπτώσεων της μεγαλύτερης αστάθειας για ε, που προκαλείται από την ε, ε οικονομία. Ε, Όλα αυτά οδήγησαν στην εξαφάνιση της πίστοσης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί μια τράπεζα η οποία είναι συγκεντρωμένη και είναι προσανατολισμένη όλο ένα και περισσότερο στις πολυεθνικές εταιρείες και στην ε, κερδοσκοπία, την χρηματιστηριακή δεν μπορεί να αναπτύξει πολιτική πιστώσεων σε ένα μικρό ε, επιχειρηματικό κύκλο. Άρα λοιπόν με αυτή την πρόταση ένωσης ε, των κεφαλαγορών ευνοούνται οι ίδιοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι που αυτή τη στιγμή αρνούνται την πίστοση, αυτοί ακριβώς δηλαδή που ασχολούνται με την κερδοσκοπία και μάλιστα μεταφέρεται ο κίνδυνος αυτών των ε, νέων μέσων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέα ρύθμιση χρηματοπιστωτική και τραπεζική με συνιστόσα δημόσια και περιφερειακή αν πραγματικά θέλουμε να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη και πρέπει μάλιστα να εμβαθύνουμε σε αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τις αρχές της τραπεζικής ε, διαχείρισης που η Κομισιόν επιμένει να αποσυνδέσει τελείως. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, ο κύριο Φιλίπ Σε Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε τι ωραία που συνεργάζονται οι Βέλγοι. Γιατί άλλοι μας κατηγορούν που δεν συνεργαζόμαστε καλά. Πάρα πολύ ωραία συνεργαζόμαστε. Θα μιλήσω αγγλικά όμως. Μας συνεργάζει πάντα να βλέπουμε το βαθμό ένταση που επικρατεί σε αυτή να βλέπουμε το αυτή την Επιτροπή όταν μιλάμε για τόσο σημαντικά θέματα. Οι μικρομεσαίες είναι πολύ σημαντικό θέμα προφανώς. Ίσως κύριε Σάιμον έχετε δίκιο ότι εδώ και 20 χρόνια βασικά ε, ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Να πω ότι ίσως για πρώτη φορά θα διαφωνήσω ελαφρώς μαζί σας. Όταν διαβάσει κανεί τα τελευταία έκθεση τη ΕΚΤ για, πρόσβαση στη, για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και σας παραθέτω λέει οι μικρομεσαίες τη ευρωζώνη θεωρούν πως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι το λιγότερο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. <laughs> Εγώ δεν είμαι απόλυτος ε, τυφλός πιστός της ΕΚΤ, αλλά αν αυτό είναι πραγματικότητα, μάλλον υπάρχουν και άλλα προβλήματα σημαντικά που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η ζήτηση για τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους, η εξασφάλιση της ζήτησης είναι το πιο σημαντικό που τους απασχολεί. Γι' αυτό κάπως δεν αισθανόμαστε πολύ άνετα με αυτή, τη, με αυτή την ε, πρόταση, ότι δηλαδή θα πρέπει να χαλαρώσουν οι προληπτικοί κανόνες, οι μακροπροληπτικοί κανόνες για να μπορέσει να προωθηθεί η χρηματοδότηση. Θυμάστε, ε, όταν είπαμε να εξετάσουμε την Τραπεζική Ένωση να δούμε όχι μόνο μία κατηγορία, γιατί υπάρχουν διάφορα επιχειρηματικά πρότυπα στις τράπεζες και κάποιες τράπεζες κάνουν ένα, ένα πράγμα, δηλαδή χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Ορισμένες εξ αυτών μάλιστα χρηματοδοτούν αποκλειστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ξέρω κάποιες, ε, CPH ή τριώτους στο Βέλγιο, τράπεζε που χρηματοδοτούν μόνο και αποκλειστικά μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να σχεδιάσουμε με τέτοιο τρόπο τον κανονισμό τον μακροπροληπτικό, σύμφωνα, δηλαδή με τα επιχειρηματικά πρότυπα και όχι σύμφωνα με το ποιον δανείζουν. Αυτό θα σήμαινε βέβαια το να συντάξω μια CDR 5 αλλά το να χαλαρώσουμε τον κίνδυνο, τον παράγοντα κινδύνου που συνδέεται με τις ΜΜΕ θα ήταν κάπως ε, ε, κίνδυνο. Το ίδιο με την ε, τυφλοποίηση. Το συζητήσαμε με το... Αυτή η τιτλοποίηση δεν προορίζεται για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι κάτι που καθιστά ευκολότερη τη χρηματοδότηση για τις μεγάλες εταιρείες. Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα εδώ. Αυτό που εμείς θα προτείναμε και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το αναφέρουμε στην έκθεση ε, στην επόμενη γύρο του κανονισμού για τις τράπεζες, μήπως θα μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε τους μακροπροληπτικούς κανόνες, όχι σύμφωνα με τον πελάτη, αλλά σύμφωνα με το επιχειρηματικό πρότυπο. Επίσης, ε, διαπιστώνω, όταν μιλάμε στην Τραπεζική Ένωση για συμβολή στο Ταμείο Εξυγίανσης ή Καθάρισης ή στο Ταμείο Εγγύσης Καταθέσεων είναι κάτι το οποίο έχουν αντιμετωπίσει οι βελγικές τράπεζες, ότι δηλαδή οι συμβολές των τραπεζών που δανείζουν τις μικρομεσαίες, αυτές τις κοινέ τράπεζες, που στην ουσία είναι ε, α, τράπεζες αμοιβαίου κεφαλαίου για να καλύπτουν όλες αυτές, είναι δυσανάλογα ψηλό. Δηλαδή η BNP Paribas πληρώνει πολύ λίγα, σε σχέση με το σύστημά της, ενώ η Ρεμπέκα Φανμπρέντα χρησιμοποιεί ένα πολύ μεγάλο ποσό ανάλογα με το πόσα χρήματα έχει στη διάθεσή της, τα κεφάλαιά της. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε κάπως να διευκολύνουμε αυτές τις τράπεζες, να είμαστε λίγο πιο δίκαιοι. Επίσης ένα θέμα το οποίο ε, σιγοπεθαίνει, αργοπεθαίνει είναι εκείνες οι τράπεζες ε, ε, που ασχολούνται με την κερδοσκοπία. Να τους πούμε ότι σε αυτές τις τράπεζες έχουμε κλείσει τις πόρτες του καζίνου. Άρα πρέπει να στραφούν στην πραγματική οικονομία και να επανέλθουν στις επενδύσεις. Και κάτι ακόμα, πάντως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι να αναζωογονήσουμε γενικώ το μακροοικονομικό περιβάλλον. Και γνωρίζω ότι έχουμε το εφσί αλλά θα έλεγα ότι είναι μικροσκοπικό. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει κάποια στρατηγική κατεύθυνση. Πιστεύω πως εάν στοχεύσουμε τις δημόσιες επενδύσεις και φυσικά μιλώ για την ενεργειακή μετάβαση που είναι ένας τομέας όπου πολλές μικρομεσαίες έχουν να παίξουν ρόλο αντί για πυρηνικά εργοστάσια γιατί μιλάμε εδώ για ηλιακή, αιωλική ενέργεια. Αυτά είναι για τις μικρομεσαίες Εάν λοιπόν η ενεργειακή μετάβαση μετατραπεί στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Επενδύσεων. Αυτό θα βοηθήσει πολύ όλες τις μικρομεσαίες, αυτά, αλλά αυτό δεν είναι θέμα αυτής της συνομοθεσίας. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ, Διευθυντή, ο κύριος Τζάνι. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπα πέντε προηγουμένως γιατί νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Όποια στατιστική και αν εξετάσουμε, όποια και αν έρευνα να κάνουμε ανάμεσα στις μικρομεσαίες και στις, στους επιχειρηματίες, σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν το τι ανάγκη έχει η πραγματική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο θέμα το οποίο πάντα θέτουν, η πρώτη τους ανησυχία, δεν είναι η απλή πρόσβαση στην πίστοση. Είναι κάτι το οποίο έχει πράγματι βελτιωθεί τον τελευταίο καιρό, αλλά η έλλειψη ζήτησης για τα προϊόντα τα οποία παραγούν. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να δώσει εγγυήσει για μια ουσιαστική ζήτηση και τόνωση της ζήτησης, τότε οι μικρομεσαίες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να πτωχεύουν. Αν ακολουθήσουμε την ίδια κατεύθυνση, που ακολουθήσαμε σε επίπεδο μακροοικονομικό μέχρι τώρα, μέσω της επιβολής της λιτότητας, μέσω της επιμονής σε επίπεδο διαθρωτικών αλλαγών, τότε οι ανησυχίες των μικρομεσαίων δεν θα καλυφθούν ποτέ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και ένα άλλο θέμα το οποίο αποτελεί μια μεγάλη δυσκολία για τις μικρομεσαίες είναι το θέμα του ενιαίου νομίσματος. Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ασθενέστερων χωρών αναγκάζονται να λειτουργούν κάτω από συνθήκες χειρότερες από τις μικρομεσαίες των ισχυρών. Για ποιο λόγο? Γιατί οι περιφερικές μικρομεσαίες στην ουρχία έχουν μια συναλλαγματική ισοτιμία υποτιμημένη σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τους και αυτό είναι ένα τρομακτικό θέμα. Τώρα, αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να περιλαμβάνετε στην έκθεσή σας θα ήταν να προσπαθήσετε να συγκεντρώσετε την προσοχή σας και στο θέμα της πρόσβασης στην λεγόμενη παραδοσιακή πίστοση. Οι αγορές κεφαλαίων φυσικά δεν είναι φτιαγμένες ε, για τις μικρομεσαίες. Ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να λειτουργεί στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου το μέσο μέγεθος μιας επιχείρησης είναι πολύ μεγαλύτερο από μια ευρωπαϊκή το σύστημα αυτό δεν ισχύει στην Ευρώπη. Η αγορά των κεφαλαίων και ε, τα ομόλογα, οι τιτλοποιήσεις δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για τις μικρομεσαίες, αλλά μόνο για τις μεσαίες και μεγάλες. Συνεπώς λοιπόν ε, νομίζω ότι εδώ κάνουμε προσπάθειες οι οποίες δεν θα αποδώσουν τίποτα. Ας συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στον τραπεζικό τομέα. Ο τραπεζικός τομέας στο μέλλον θα είναι ο βασικός τρόπος πρόσβασης στην πίστοση των μικρομεσαίων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να κάνουμε το εξής. Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει ένα σύστημα πιστοτικό το οποίο να συγκεντρώσει την προσοχή του στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή να παίξει έναν ρόλο δημόσιο να εγγυάται την πρόσβαση στην πίστοση των μικρομεσαίων. Ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα πιστοτικά ιδρύματα. Υπάρχουν πάρα πολλές τράπεζες στην Ευρώπη, υπάρχουν πολλές μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη, οι οποίες αφιερώνουν ε, τον προϋπολογισμό τους, το μέγιστο τμήμα του, σε δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική οικονομία. Και αυτό δεν δημιουργεί αξία για την οικονομία, δεν υποστηρίζει την οικονομία, δεν υποστηρίζει τις μικρομεσαίες, υποστηρίζει όμως την καταχρηστική, ε, μια καταχρηστική μορφή επενδύσεων και δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους στο εσωτερικό της Ένωσης με κινδύνους μιας νέας κρίσης χρηματοπιστωτικής ή βάρος πάντα των μικρομεσαίων. Την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα εξαιρετικό άρθρο το είπε και ο υπεύθυνο της ΦΕΔ ε, στη Μινεάπολη, ο οποίος ήταν και ένας από τους υπευθύνου της πολιτικής που έσωσε τις μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις μετά την κρίση του 2008 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική ανακατανομή των τραπεζών στην Ευρώπη έτσι ώστε κάποιες από αυτές να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, γιατί οι υπόλοιπες δραστηριότητες υπιστοτικές δεν μας αφορούν. Κατά τα άλλα τώρα υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία στην έκθεση, το λεγόμενο peer-to-peer -peer ε, lending, δηλαδή η έλλειψη ενδιαμέσου είναι ένα μέσο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε τους κανόνες που ισχύουν έτσι ώστε να διευκολύνουμε για τις μικρομεσαίες την πρόσβαση σε αυτό το μέσο το οποίο βοηθά στη χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών που από τα παραδοσιακά κανάλια δεν θα μπορούσαν να βρουν χρήματα. Ένας άλλος τομέας θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης venture capital δημόσια τα οποία να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις καινοτόμες επαναλαμβάνω οι οποίες στον ιδιωτικό πιστοτικό τομέα δεν θα βρουν βάσεις χρηματοδοτικές και δεν θα χρηματοδοτηθούν από τις μεγάλες τράπεζες, αλλά επιχειρήσεις οι οποίες ε, προοπτικά θα προσφέρουν τη θέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νέες τεχνολογίες, νέα επιχειρηματικά πρότυπα, νέες μελλοντικές προοπτικές. Αυτές οι ιδέες ε, δεν ε, προσφέρουν άμεση απόσβεση και απαιτούν υψηλές επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και υποδομές. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε έτσι ώστε ο τομέας ο δημόσιος και αυτός να συνεισφέρει στη στήριξη των καινοτόμων ιδεών που θα δημιουργήσει επιπλέον κέρδη για την πραγματική οικονομία. Ένα τελευταίο σημείο. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με την έκθεση αλλά έχει μεγάλη σημασία και αυτό Νομίζω ότι έχουμε ένα μειονέκτημα σαν μικρομεσαίες σε σχέση με τις μεγάλες. Είναι το θέμα της φορολογίας. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και το είδαμε αυτό και στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής Τάξ και στα πλαίσια των εργασιών της δικής μας Επιτροπής για την φορολογία των επιχειρήσεων. Έχουν ειδικέ ευνοϊκές μορφές φορολογίας οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό συνιστά σαφέστατα μια στρέβλωση της αγοράς την οποία υφίστανται τις συνέπειες της εννοώ οι μικρομεσαίες. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ισότητας ανάμεσα στις μικρές και μεγάλες και στον φορολογικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο τώρα, ένα τέταρτο για το λεγόμενο catch the eye. Δεν ξέρω όμως αν κάποιος θα ήθελε το λόγο. Το θέμα είναι σημαντικό. Uh, the floor to Ο κύριος Καράς έχει τελικά το λόγο. Σας ευχαριστώ για τα θέματα και για τη συζήτηση αυτή, αυτή για τέτοια θέματα σημαντικά. Και για τη λεπτομερή αυτή τη συζήτηση. Και έχω να πω ότι κάθε παρέμβαση είχε και περιλάμβανε ένα γενικό τμήμα το οποίο ξεπερνά τα όρια της έκθεσης αυτής και κάθε παρέμβαση είχε και ένα συγκεκριμένο τμήμα για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και να συμπληρώσουμε την έκθεση αυτή. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να επισημάνω ένα στοιχείο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια τα πλαίσια της ρύθμισης των τραπεζών συνέβησαν πολλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είμαστε στο μηδέν. Χωρίς το κοινοβούλιο μας δεν θα υπήρχε το supporting factor. Χωρίς το κοινοβούλιο δεν θα υπήρχε... Δεν θα υπήρχαν ε, υποχρεώσεις ε, για τις αποκεντρωμένες τράπεζες, για την ενίσχυση των αποκεντρωμένων τραπεζών. Χωρίς το κοινοβούλιο στο ΕΦΣΙ δεν θα υπήρχε ενίσχυση των promotional banks. Δεν θα υπήρχε ξεχωριστό μερίδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν θα υπήρχε σχέδιο επενδύσεων χρειάζεται μια αξιολόγηση των όσων έχουν συμβεί βάσει των υφιστάμενων και των ε, παλαιών εκθέσεων. Σύμφωνοι, δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε όλα, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα επαναλάβουμε. Και φυσικά θα πρέπει να κάτσουμε και να ελέγξουμε ποιες ήταν οι συνέπειες του χρηματοοικονομικού κανονισμού σε ό,τι αφορά την εχώρηση τέτοιων χρηματοδοτικών μέσων προς τις τράπεζες. Ασφαλώς. Αλλά στην έκθεση πρωτοβουλίας αυτή το θέμα είναι... Το θέμα μάλλον δεν είναι να καταρτήσουμε μια έκθεση για τις τράπεζες, ούτε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση του τραπεζικού κλάδου. Δεν έχουμε εκθέσεις άλλες. Αλλά έχουμε και μια ξεχωριστή ε, έκθεση σε ό,τι αφορά την τυπλοποίηση για τις κεφαλαγορές. Θα πρέπει να πούμε ποιος είναι ο δρόμος για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις κεφαλαγορές. Δεν έχει νόημα να μετατοπίσουμε όλη τον τομέα χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από, τον, από τα δάνεια στι κεφαλαγορέ. Το είπαν πολλοί συνάδελφοι θα πρέπει να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε την χορηγήση δανείων. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το πώς ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης, γιατί με την έκθεση αυτή δεν μπορούμε να καθορίσουμε την φορολογική και οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι θέμα διαφορετικών αρμοδιοτήτων. Και ως εκ τούτου θα ήθελα να σας παρακαλέσω στις τροπολογίες που θα καταθέσετε να έχετε ως σκοπό βασικά το να συμπληρώσετε την έκθεση προκειμένου και το συντομότερο δυνατόν να κάτσουμε να συζητήσουμε σε μια συνάντηση των σκιωδών ποια θα είναι τα σημεία στα οποία θα δώσουμε βάρος στην έκθεση. Εγώ προσπάθησα αφενός να ορίσω τη χρηματοδότηση μέχρι δανείων ως ένα τμήμα της χρηματοδότησης, όχι 100% και το θέμα των startups, των νεοφιών, ε, των promotional banks, ε, των crowdfunding, να τα περιγράψω ως κάτι συμπληρωματικό και να θέσω στο επίκεντρο απλοποιημένες ρυθμίσεις. Γιατί προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να κινηθούμε, θεωρώ. Όχι είτε το ένα είτε το άλλο, διαζευκτικά, αλλά διεύρυνση του χρηματοδοτικού πλαισίου και συμπερίληψη όλων αυτών των μέσων. Αν όλοι πιστεύουμε ότι το θέμα της χρηματοδότησης δεν αποτελεί ένα πρόβλημα, αλλά ότι μόνο το θέμα της ανταγωνιστικής πολιτικής και το θέμα της ανάπτυξης είναι αυτό που μας απασχολεί, θα πρέπει αυτό να μπει στην έκθεση. Γιατί με την έκθεση αυτή δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα που άπτονται της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής ανάπτυξης. Γιατί άμα θέλουμε να πούμε ότι δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε καν το θέμα τη χρηματοδότηση, γιατί δεν αποτελεί πρόβλημα, ε, μην κάνουμε την έκθεση. Αν πούμε ότι έχουμε ένα θέμα ανταγωνισμού, ανάπτυξης, πρόσβασης, θα συμφωνήσω. Απλά πιστεύω ότι καλό είναι να υπάρχει και μια πολιτική για τη χρηματοδότηση. Και ο συνάδελφος από τους Σελδημοκράτες το είπε αυτό και το έθεσε πάρα πολύ ορθά. Είπε και μίλησε για παραδείγματα τα οποία στον Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν πολύ πιο άσχημα από ό,τι σε άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το θέσουμε και αυτό το θέμα και θα πρέπει αυτή η έκθεση να αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Κεφαλαγορά. Uh, Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τον κύριο Κάρασα. Και έτσι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και τώρα ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 2, για τις ε, απαλλαγές σε ό,τι αφορά τους εμπόρους ε, τέτοιων προϊόντων. Εγώ είμαι ο συγητής. Να σας πω ότι το CRR εξαιρεί στην παρούσα φάση τους εμπόρους αυτούς από τις σχετικές απαιτήσει και οι δύο αυτές ε, έτσι θα υπάρξει χρόνος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μια αναθεώρηση του προληπτικού καθεστώτος που εφαρμόζεται και εφόσον κρυθεί κατάλληλο να υπάρξουν ε, επίσης ε, διαφορετικές προτάσεις και για το προφίλ κινδύνου, τα προφίλ κινδύνου των εμπορευομένων σε βασικά προϊόντα. πιθανές αλλαγές στην παρούσα φάση ε, ε, δεν έχουν οριστικοποιηθεί. αλλά θα πρέπει οι διαδικασίες όλες αυτές να ολοκληρωθούν, όποια από τις δύο ολοκληρωθεί πρώτα μέχρι τις αρχές του 2020. Ιδιαίτερα σε σχέση ε, με το πέρασμα στο νέο καθεστώς μετά από δύο ή τρία χρόνια. Εμείς συμφωνούμε λοιπόν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίνουμε ε, την ε, ε, παράταση. I just Μόλις ονοκλήρωσα. Είναι τεχνικό το θέμα, είναι εύκολο ως εκ τούτου. Ζητώ συγγνώμη από, από τη διευμηνία γιατί δεν ακούγεται αυτό το οποίο λέω. Τώρα για τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Μπάλτς. Thank you very much, uh, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλια που κάνετε. Η κυρία Πιετικά είναι συμφωνή με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την οποία άλλωστε υποστηρίζει και ο εισηγητής. Θα ήθελε ωστόσο να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της για τις επενδυτικές ε, επιχειρήσεις και να βρει μία προσέγγιση η οποία θα συμφωνηθεί στην παρούσα φάση και περίοδο εξαιρέσεων και απαλλαγής. Γιατί είναι σαφές ε, ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο για τους εμπόρους αυτούς. Η κυρία κάνει λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, τις, να διευκρινίσει κατά πόσον με την αναθεώρηση αυτή έχουν ήδη κάποια σχέδια και κάποιο χρονοδιάγραμμα κατά νου για την υποβολή των προτάσεών τους. Αυτά ήταν τα σχόλια από πλευράς της κυρίας Πιελικάνιν που είναι σκιώτης από πλευράς του ΕΛΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπάλτ. Θα σε ευχαριστούμε τώρα από την Άλντε ο κύριος Τόιρερ. ευχαριστώ στην Άλντε. σύμφωνη, η Άλντε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει αυτή η απαλλαγή σε ό,τι αφορά στους διαπραγματευτές της εγγραμματιστρία βασικών ευμαρμάτων. Όπως βλέπετε από το σχετικό κανονισμό, ιδάλλως ε, οι απαλλαγές αυτές θα εκπνεύσουν του Δεκέμβρη του 17 και οι διαπραγματευτέ αυτές θα υπόκεινται σε όλες τις σχετικέ υποχρέωσει. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αποτελούσε την πιο σωστή αντιμετώπιση και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε τομεί όπου οι διαπραγματευτέ αυτέ δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα, όπω στην ενέργεια και στην γεωργία. Γιατί το προφίλ σε ό,τι αφορά το ρίσκο αποτυπώνει την κατάσταση στην αγορά. Υπάρχει λοιπόν μια φυσική έκθεση των εταιριών αυτών. Έχει να κάνει και με την ζήτηση, την φυσική ικανότητα και ούτω καθεξής δεν εξαρτώνται πάρα πολύ από την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Ωστόσο, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εντέλεχο τη φύση και το ρίσκο που αναλαμβάνουν σχετικέ εταιρείε σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του καθεστώτο για τι κεφαλογικέ απαιτήσει προκειμένου να υπάρξει και να διαμορφωθεί το σωστό νομοθετικό πλαίσιο. Thank you, Mr. For the Group, uh, Madame Mattia. κυρία Ματίας από την ΚΟΕ. So we go to, uh... Ναι, είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Λάμπερτς από τους Πράσινους και έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τους πολιτικούς συνήθως είναι να καταφέρουν να μην μακρηγορήσουν. Εγώ το αντίθετο έχω να αντιμετωπίσω σήμερα. Δεν θέλετε να μακρηγορήσω ασφαλώς για το δύσκολο αυτό το θέμα. Συμφωνούμε λοιπόν με τον εισηγητή. Αλλά μια και έχω ακόμα χρόνο ομιλίας, να σας πω ότι από το Σάββατο έγινε και παππού πρώτη φορά. Για να ελαφρώσουμε κάπως την ατμόσφαιρα. Εγώ ότι δεν έκανα τίποτα, η κόρη μου. Τα κατάφερα. Πέραν αυτού όμω, ε, τι να σα πω, υποστηρίζουμε τον εισηγητή. Ε, Εξαιρετικά. Η FTD, ENF, δεν βλέπω να θέλετε το λόγο. Μάλιστα. 21 ημερολογικέ μέρε για να υποβάλλετε αντιρρήσει στο φάκελο. Αυτό μέχρι 7 Μαρτίου. Μετά από την ημερομηνία αυτή θα θεωρηθεί εγκεκριμένη η έκθεση αυτή εκτός και αν 10% υποβάλλει ένσταση 7 μέλη, δηλαδή της Επιτροπής μας. Και έτσι ολοκληρώσουμε και το σημείο αυτό και θα ήθελα να επανέλθω στο προηγούμενο σημείο που ξέχασα να σας πω ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα για την προηγούμενη έκθεση. Για την έκθεση επαναλαμβάνω για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. 5 Απριλίου Προθεσμία για τροπολογίε 12 ε, το μεσημέρι. Εξέταση των ε, τροπολογιών 25-26 Απριλίου. ...25 26 Απριλίου. Η ψηφοφορία στις 13 ή 14 Ιουνίου στην Επιτροπή Οίκων. Και την Ολομέλεια το Σεπτέμβριο, με το καλό. Και έτσι περνάμε στο τελευταίο σημείο της ε, σημερινής συνεδρίασης μας. Πρόεδρε, κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η διερμηνία γιατί το μικρόφωνο σας δεν λειτουργεί. Ίσως θα μπορούσατε να το φροντίσετε να το φροντίσουν οι τεχνικοί, εν περιπτώσει. Otherwise, ε, Ή να χρησιμοποιήσετε το διπλανό μικρόφωνο. But so for the timetable... Ε, Για τις μικρομεσαίες, λοιπόν, προθεσμία για τις τροπολογίες 5 Απριλίου, εξέταση 25 και 26 Απριλίου, 13 και 14 Ιουνίου ψηφοφορία στην εικόνα και είπαμε με το καλό στο, στην Ολομέλεια θα πάτε το Σεπτέμβριο και έτσι περνάμε στο τελευταίο ζήτημα, στο τελευταίο θέμα μάλλον της σημερινής ημέρης της διάταξης, ναι, ναι, ναι, στο θέμα για το ΦΠΑ. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Κοινό σύστημα ΦΠΑ. Η κυρία Φερέρα. Thank you very much. I'll do that. ευχαριστώ. Θα το παρουσιάσω αυτό λόγω του, στη θέση του Πέτε Ζήμεν, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν για πολύ σοβαρου λόγου. Ο κ. Πετεζήμων πιστεύει ότι η έκθεση είναι μια τεχνική πρόταση ουσιαστικά για την παράταση του ελάχιστου συντελεστή του 15% από την 1η Ιανουαρίου 16 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 17. Η οδηγία αυτή είναι στην ουσία το μεταβατικό σύστημα ελαχίστου συντελεστού. Δεν θα πρέπει να υπάρξει κατώτερο ποσοστό συντελεστού κάτω από το 15% σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Το ελάχιστο αυτό ποσοστό νομίζω ότι είναι ε, ε, μια σωστή, αν θέλετε, ρήτρα ασφαλείας για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Όσο για τις χώρες που έχουν κατώτερο κάτω του 15%, οι υπάρχουσες ρυθμίσεις δημιουργούν το περιθώριο για τα κράτη-μέλη να επιτρέπουν την επιστροφή ΦΠΑ έτσι ώστε ε, να υπάρχει αν θέλετε μια κάποια εξίσωση μέσω της μείωσης ουσιαστικά του φόρου. Η παράταση αυτή δεν είναι η πρώτη, πέντε φορές έχει ισχύσει και όπως είπα έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2015. Το 2016 φέτος δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα τελικό σύστημα, μια πρόταση τελικού συστήματος ασφαλούς που δεν θα προσφέρεται σε φαλκιδεύσεις. Μετά από τα επιτεύγματα θα έλεγα στα οποία καταλήξαμε στη συνέχεια της ανακοίνωσης του 2011 ε, για τις μελλοντικές μορφές ΦΠΑ. Για το εμβοκινοτικό εμπόριο λοιπόν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφείς όπως και οι προτάσεις για μεταρρυθμίσεις σε σχέση με την αλλαγή των κανόνων για, τις, για τα ενδιάμεσα επίπεδα συντελεστών. Το τελικό, η τελική μορφή και το τελικό καθεστώς θα γίνει μέσω της πρότασης, καθοριστεί μέσω της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το 15%. Προς το παρόν λοιπόν είπαμε ε, θα ισχύσει η πρόταση αυτή ε, μεταβατικά μέχρι το τέλος του 2017 και θα περιμένουμε το επόμενο πρόγραμμα δράσης, δεν θα σας κουράσω άλλο. Thank ε, Ευχαριστώ Ελίσα η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν είναι παρούσα, αλλά έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Λάγκεν. Uh, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Επί θα αρχής ασφαλώς συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Είναι διαδικασία συνένεση. Θα πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση, αλλά εδώ πέρα έχουμε κάποιε ιδιαιτερότητε, κάποια παράξενα πράγματα. Το πρώτο παράξενο είναι γιατί είναι η παράταση για δύο έτη μόνο, έως το έκανε πέντε χρόνια. Δεύτερο παράξενο. Και εδώ πραγματικά ανακύπτει το ερώτημα του πού οφείλεται μεταξύ 1η Ιανουαρίου και 1η Απριλίου που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τι θα γίνει, θα πρέπει να πληρώσουμε μέχρι την Ολομέλεια, θα υπάρχει τρει μήνε ένα κενό νομοθετικό. Δεν θα υπάρχει νομοθεσία. Η νομοθεσία ε, σταμάτησε να ισχύει το Δεκέμβριο του 2015. Γιατί καθυστέρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο και γιατί μόνο για δύο χρόνια είναι αυτή η πρόταση και γιατί με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Όλοι λένε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την απάθεια στο ΦΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει έτσι τρει μήνε να περάσουν. Είναι ανεξήγητο. Και θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή αυτό κάπου να το επισημάνουμε στην έκθεση. Εγώ στο λιγότερο το βρίσκω αυτό περίεργο. Ε, thank you, Mr. Langen. Σας ευχαριστούμε κύριε Λάγκεν. Για το ECR είμαι εγώ ο σκιώδης εισηγητής. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Σίμων. Συμφωνήσαμε δε με τον ε, ε, εισηγητή και την Επίτροπο και την Επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρξει παράταση δύο ετών. Ελπίζουμε μέσω προσύνη να αξιοποιήσει το χρονικό διάστημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταρτήσει ένα σωστό σχέδιο δράσης για το ΦΠΑ και προκειμένου να καταστήσει η διασυνοριακή συναλλαγή κάτι πιο απλό για τις ε, μικρομεσαίες, γιατί δυστυχώ συχνά ακόμα λαμβάνουμε καταγγελίε από μικρομεσαίε επιχειρήσει για το καθεστώ του ΦΠΑ. Είναι πολύ βαρύ, δυσκίνητο, δυσκολία ανάκτηση του ΦΠΑ από άλλε. Ε, χώρες προβλήματα για τις ε, ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Άρα ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εστιαστεί μόνο στην καταπολέμηση της απάτης, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να ολοκληρώσουμε και αυτή την ενιαία αγορά. Να ανοίξουν νέε πόρτε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει με ένα πιο απλοποιημένο καθεστώ ΦΠΑ. Συμφωνώ όμω και με τον κύριο Λάγκεν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει κάποια απάντηση να δώσει, αλλά πραγματικά ελπίζω τα δύο χρόνια να τα χρησιμοποιήσει και να τα αξιοποιήσει για να προτείνει κάτι πιο σωστό. Από την άλλη, τώρα ο κύριος Γέσεκ ε, έφυγε. Από τους πράσινους ο κύριος Ουρθάσου και αυτός αποχώρησε. Και έτσι έχουμε και λίγο χρόνο για κάτι Η FTD, η NF. No. Anyone uh, still Άλλος κανείς στη δικασία Catch the ή δάλλως μπορούμε να ολοκληρώσουμε λίγο πιο νωρίς τη σημερινή μας συνεδρίαση. Το χρονοδιάγραμμα και να πάρει το λόγο η κυρία Φερέρα από πλευράς του εισηγητή. You Well, thank you very much. I think there is no... Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Είναι σημαντικό ωστόσο να κατανοήσουμε από την Κομισιόν και εδώ επιβεβαιώνω αυτή την αίσθηση που παρουσίασε ο κύριος, Βαντε, ο κύριος Λάγκε, ο κύριος μάλλον, ότι έτσι πολύ αργά πήραμε την πρόταση και ότι Θεωρήσαμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα, τα δύο χρόνια, χρειάζονταν για να, ολοκληρώσει, να ολοκληρωθεί μια ευρύτερη μεταρρύθμιση της λειτουργίας του ΦΠΑ και γνωρίζουμε ότι στην ΕΚΟΝ παρακολουθούμε πολύ στενά ε, τα θέματα της καταπολέμησης απάτης σε σχέση με το ΦΠΑ. Φυσικά θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε την Επιτροπή και να επιβεβαιώσουμε το κατά πόσο το ερμηνεύουμε όλα αυτά με το σωστό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Μόλις ε, μου είπαν ότι η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη την ερώτηση, θα εξετάσει το θέμα και θα επιβεβαιώσει εάν αυτό συνδέεται με την ευρύτερη ε, μεταρρύθμιση ΦΠΑ ή όχι. Άρα λοιπόν ε, το επεισόδιο έχει συνέχεια. Έχουμε λοιπόν το θέμα αυτό υπό την απλοποιημένη δικασία, οπότε έχουμε 25 μέρες να ε, υποβάλουμε τις αντιρρήσεις μας, δηλαδή μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα θεωρηθεί πως εγκρίνεται η έκθεση. Και έτσι εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.